Εντάξει είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους Ερωτές Σώματος και δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο των στρατηγικών κατά της τρομοκρατίας. Εξ του Συμβουλίου, για να αρχίσει τη συζήτηση, ο κ. Πέρες Ρουμπαλκάμπα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την παρέμβασή μου σε αυτή τη συζήτηση ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που προσφέρεται να διεξαχθεί μια τέτοια συζήτηση για το ότι μπορούμε να συζητήσουμε uh, Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για έναν πρόεδρο είναι πώς να είναι αυστηρός με τους αρχηγούς των ομάδων αλλά πρέπει να το κάνω κύριε Σούλτς παρακαλώ κύριε Κονπεντίτ, κύριε Φερχόφστατ μιλάει το Συμβούλιο εδώ πέρα γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε τις ιδιωτικές σας συζητήσεις αλλού ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σας έλεγα ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωβουλή για τη δυνατότητα που υπάρχει να διεξαχθεί μια ήρεμη νυφάλια συζήτηση για τα θέματα της τρομοκρατίας και κάποια από τα στοιχεία της πολιτικής κατά της τρομοκρατίας συγκεκριμένα. Και αυτό σε σχέση με τα όσα ε, δημιουργήθηκαν μετά το, την απόπειρα στο Detroit ε, και την συναισθηματική φόρτιση όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι κατανοητό αυτό, αλλά είμαι υπέρ του να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να εργαστούμε με συνεχή, συνεκτικό τρόπο, χωρίς βιασύνη, αλλά και χωρίς καθυστέρηση, όταν έχουμε μια τέτοια απειλή μπροστά μας, σαν την απειλή της τρομοκρατίας, που πρέπει να πω ενώπιον των Ευρωβουλευτών, δεν μειώθηκε καθόλου η διάσταση αυτής της απειλής όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες μας. Ξέρουμε ότι μας παρατηρούν οι τρομοκράτες ε, και ξέρουμε ότι προσπαθούν να αλλάξουν μορφές δραστηριοποίησης και θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε στρατηγικές αποτελεσματικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και γι' αυτό αυτή η στρατηγική πρέπει να έχει καινοτόμο χαρακτήρα και να βελτιώνεται και να αλλάζει και πρέπει κυρίως να μαθαίνει από τα λάθη από τα όσα λάθη κάνουμε στο παρελθόν, ε, κάναμε στο παρελθόν. Τούτων λεχθέντων είναι προφανές ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αποτυχημένη απόπειρα το Δεκέμβριο στο Ντιτρόιντ, αυτή τη στιγμή δεν θα το συζητούσαμε αυτό το θέμα υπό αυτού του όρου. Δηλαδή, στην ουσία αυτή τη συζήτηση βρίσκεται μια ολόκληρη σειρά προληπτικών δράσεων και συμπερασμάτων και στρατηγικών που απορρέουν από την ανάλυση αυτών των γεγονότων, όπως για παράδειγμα αυτού του Detroit, στο οποίο αναφέρθηκα. Στην ουσία αυτής της συζήτησης βρίσκεται η ανάλυση για το τι πήγε στραβά και απέτυχε σε σχέση με αυτή την απόπειρα στο Detroit και σε σχέση με τα μέτρα που τα διαφορετικά μας κράτη υιοθετούν ώστε αυτά τα σφάλματα και τα λάθη να μην επαναληφθούν. Και γι' αυτό κάνουμε λόγο για ανάλυση στοιχείων και δεδομένων. Και γι' αυτό κάνουμε λόγο για τις υπηρεσίες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τη κοινή ανάλυσης των δεδομένων που έχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Και γι' αυτό κάνουμε λόγο και για τους προσωπικούς σαρωτές. Κάνουμε λόγο για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν σε μία απόπειρα που ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί και δεν θα επαναληφθούν τέτοια ασφάλματα. Και για αυτή τη συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν τα πιο σαφή συμπεράσματα που μπορούμε να συναγάγουμε από την αποτυχημένη αυτή απόπειρα του Detroit. Είναι πέντε αυτά τα στοιχεία. Πρώτο στοιχείο το Detroit καταδεικνύει ότι η πολιτική αεροπορία εξακολουθεί να είναι ένα αντικείμενο πρωταρχικής σημασίας ως στόχος για τους τρομοκράτες. Δεύτερο, το Detroit αποδεικνύει ότι είναι σημαντικό να συλλέγουμε στοιχεία. Όμως είναι πολύ πιο σημαντικό να εντάσσουμε αυτά τα στοιχεία και να τα αναλύουμε σε μια σωστή βάση δεδομένων. Το τρίτο στοιχείο αποδεικνύει το Detroit ότι οι διάφορες υπηρεσίες της Αλκάιντα είναι σε θέση να μπορούν να δράσουν εκτός του, της δικής τους περιφέρειας. Το ίδιο για παράδειγμα όσον αφορά την Αλκάιντα της Χερσονήσου, της Αραβικής Χερσονήσου που βρίσκεται πίσω από τέτοια, τέτοιες απόπειρες ή ακόμα και την Αλκάιντα στο Μαγρέμπ, Ισλαμικό Μαγρέμπ. Είναι μια απειλή την οποία έχουμε ενώπιόν μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τέταρτον, μας υπενθυμίζει το Detroit τη σημασία που έχει να εργαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης την ίδια την προσωπικότητα αυτών των τρομοκρατών και η προσωπικότητα που έχει μεγάλη σημασία και μας ε, κάνει τον Detroit να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις αποτυχημένες χώρες, τα κράτη που έχουν καταρρεύσει και που αποτελούν ας το πω έτσι έναυσμα αυτών. Πρώτο και δεύτερο συμπέρασμα, ο κίνδυνος για την πολιτική αεροπορία από αυτές τις δράσεις και η ανάγκη να εντάσσουμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε σε σωστές βάσεις και ανάλυση αυτό οδηγεί στη συζήτηση άμεσα αυτών των θεμάτων απόψε ή των δύο θεμάτων που συζητούμε για την ε, πληροφόρηση και την χρήση της, πληροφορίες και τη χρήση τους και για τους προσωπικούς αρωτές σώματος. Δεν είναι η ε, μόνη φορά όπως για τον, την τελευταία έκθεση για τον συντονιστή, του συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εδώ στην Ευρωβουλή πέρυσι μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική έκθεση όπου γινόταν λόγος για την διαχείριση των πληροφοριών και των στοιχείων, των δεδομένων, καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διότι πραγματικά η πληροφόρηση και η ανάλυση των πληροφοριακών αυτών στοιχείων είναι, όπως είχαμε ευκαιρία να συζητήσουμε εδώ απόψε, είναι ακρογωνιαίοι λύθοι στοιχεία θεμελιώδους σημασίας ε, για να προλάβουμε δράσεις τρομοκρατικές και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρασία. Πρέπει να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε τους τρομοκράτες. Ποιοι και πού είναι εκείνοι που θέλουν να κάνουν κάποια τέτοια απόπειρα. Να γνωρίζουμε τα όπλα που έχουν, την υποδομή που έχουν στη διάθεσή τους, να γνωρίζουμε τα συστήματα επικοινωνίας τους, όλα αυτά μέσω βάσεων δεδομένων και μέσω πηγών πηγών εξειδικευμένων που θα αντλούμε από αυτές τις στοιχεία. Και γι' αυτό, για να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και στοιχεία διαθέσιμα, πρέπει να ανταλλάσσουμε αυτά τα στοιχεία αναμεταξύ μας και πρέπει να το κάνουμε αυτό με αποτελεσματικό, επαρκή τρόπο. Πρέπει να διαχειριζόμαστε επαρκώς αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Αληθεύει και σπέβδω να το πω ότι κάποιες από τις απόπειρες που έγιναν στο παρελθόν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν οι πληροφορίες αυτές είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα εκείνων που είχαν την ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έγκαιρο, έγκαιρα όμως, με τρόπο τέτοιο που να μπορούσαν έγκαιρα να έχουν δράσει με ενσωματωμένο, ολοκληρωμένο, ευφυή τρόπο, ευφυή τρόπο. Και αυτό οδηγεί στη συζήτηση για τη διαχείριση των πληροφοριών και των δεδομένων. Για όλα αυτά, για να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρξει σωστή διαχείριση και να γίνεται επαρκώς, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση έχουμε μια στρατηγική. Μια στρατηγική που πρόσφατα εγκρίναμε. Πράγματι αποτελεί τμήμα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου από πέρσι τον Νοέμβριο που θέλει να δημιουργηθούν οι όροι και προϋποθέσεις από πλευράς των υπηρεσιών ασφάλειας των αναγκαίων εκείνων στοιχείων που μπορούν να είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα αναγκαία στοιχεία μόνο και τίποτα παραπάνω διότι η πληθώρα στοιχείων πηγαίνει ακριβώς, αντιβαίνει ακριβώς την αποτελεσματικότητα που πρέπει να διασφαλίζεται. Όπω αντανακλάται σε αυτή τη στρατηγική, αυτό που θέλουμε είναι οι αποφάσει για την ανταλλαγή πληροφοριών να γίνονται με συνεκτικό τρόπο, αποτελεσματικά, συντονισμένα, επαγγελματικά, αξιόπιστα και με αποδεκτό τρόπο για το σύνολο των πολιτών και το σύνολο των επαγγελματιών που τι χρησιμοποιούν. Μια στρατηγική αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο που πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπω επίση αντανακλάται σε πολλέ από τι δηλώσει τη Ευρωβουλή και το ψηφίσματα τη Ευρωβουλή να ανταποκρινόμαστε στι ανάγκε καταπολέμηση τη τρομοκρατία, καθώ επίση και να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα τα προσωπικά δικαιώματα των ατόμων καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Όπως σας έλεγα στην αρχική μου παρέμβαση, μεταξύ των συμπερασμάτων που μπορούμε να συναγάγουμε από την απόπειρα του Ντιτρόιτ είναι ότι τα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας εξακολουθούν να είναι πρωταρχικοί στόχοι των τρομοκρατών. Κατάφερε να, να ανέβει σε αυτό το αεροπλάνο με επαρκή ποσότητα εκρηκτικών ώστε να πυροδοτήσει αυτά τα εκρηκτικά και να εκραγεί το αεροπλάνο. Όλα τα συστήματα λοιπόν στα αεροδρόμια μας ή με άλλο τρόπο, ας το πω έτσι, είναι προφανέ ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τον εξοπλισμό ασφάλειας που έχουμε στα αεροδρόμια μας, διότι ήταν ανεπαρκής για να αποφευθεί μια τέτοια απόπειρα, που είμαστε τυχεροί που δεν συνέβη όπως συνέβη με την απόπειρα ακριβώς του Detroit που απέτυχε και δεν εξεράγει το αεροπλάνο. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε λοιπόν τις υπηρεσίες ασφάλειας και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ότι οι ύποπτοι αυτοί οι τρομοκράτες να μην μπορούν να ανεβαίνουν στα αεροπλάνα μας. Τώρα, το να ένας ο οποίος έχει όπλα ή ε, εκρηκτικά ή ε, πυροδοτικά τέτοια ε, μηχανήματα να μην μπορούν να επιβιβαστούν στα αεροπλάνα μας. Και έτσι θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρξουν τέτοιου είδους συμβάντα εν πτήση όταν το αεροπλάνο έχει απογειωθεί. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, θέματα που ανησυχούν τους ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο για, τα, για τους σαρωτές και τους body scanners, σαρωτές σώματος. Γνωρίζετε ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα για να θεσπίζει στόχους και να καθορίζει κανόνες. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών είναι εκείνο στο οποίο συζητώνται αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα της ε, ασφάλειας στα αεροπλάνα ήταν αντικείμενο στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών που έγινε πριν από κάποιες εβδομάδες στο Τολέδο. Σε αυτό το Συμβούλιο συμφωνήσαμε διάφορα πράγματα. Πρώτον, ότι είναι σκόπιμο, είναι ανάγκη να υπάρξει μια κοινή θέση στο πλαίσιο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς τους προσωπικούς αρωτέ. Γενικά για όλους τους μηχανισμούς προστασίας των αεροδρομίων μας. Δεν έχει νόημα να είναι λιγότερο προστατευμένα κάποια αεροδρόμια από άλλα γιατί τότε δεν θα είμαστε με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα προστατευόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συμφωνία με κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, είναι ένα δυσχερέ, ακαθόδε, ευαίσθητο θέμα, όπου υπάρχουν πολλέ πτυχέ που πρέπει να καλυφθούν. Πρώτη, πρωταρχικά, να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα τέτοιου είδου ε, σκάνε σαρωτών, ώστε να αποφύγουμε να επιβαστούν σε αεροπλάνα τρομοκράτε με εκρηκτικά ή τέτοια όπλα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η συμβατότητα αυτών των σαρωτών με το δίκαιο, το οποίο, τα δικαιώματα στην προσωπική ζωή και τα δεδομένα των πολιτών μας. Πράγμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο που προστατεύει η Ευρωβουλή. Και, δεύτερο, και τρίτον, να δούμε τις επιπτώσεις στην υγεία αυτών των σαρωτών για εκείνους που περνάνε από αυτούς για να επιβαστούν στα αεροπλάνα. Αυτά είναι τρία θέματα λοιπόν. Η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένα των ατομικών σαρωτών, η επιρροή τους στην υγεία και η συμβατότητα ή όχι με τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών μας Αυτά τα τρία στοιχεία, επ' αυτών των στοιχείων εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρει μελέτε που θα τεθεί στη διάθεση του Συμβουλίου και στη διάθεση τη Ευρωβουλή στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο το άτυπο Συμβούλιο ε, Υπουργών Μεταφορών στο Τολέδο αποφάσισε να υπάρξουν πρώτα αυτέ οι μελέτε για να μπορέσει να εμβαθύνει σε αυτά τα θέματα, για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε ομόφωνα σε μια θέση, κοινή θέση που θα ήταν ευκταίο να μπορέσει να επιτευχθεί. Επισημένω στο Σώμα λοιπόν ότι θα λάβουμε υπόψη το ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2008 σε μια συζήτηση που διεξήχθη για τους προσωπικούς αρωτές όπου έγινε λόγος ακριβώς για την αξιολόγηση των επιπτώσεων για τα δικαιώματα, για τις αναγκαίες διαβουλεύσεις για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις επιπτώσεις στην υγεία, για την οικονομική επίπτωση επίση και τις δαπάνες. Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική μας συζήτηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ το Σώμα για τη δυνατότητα που δόθηκε να συζητηθούν αυτά τα θέματα και ευχαριστώ Πρόεδρε για την ελαστικότητα, για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, ε, δύο επίτροποι. Πρώτα ο κύριος Κάλλας. Αγαπητοί Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Εδώ παρουσιάζουμε μια συνδυασμένη όψη ορισμένων πτυχών της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δική μου προτεραιότητα ως Επιτρόπου Μεταφορών είναι η ασφάλεια των επιβατών. Είναι τεράστια προτεραιότητα για την κοινή πολιτική μεταφορών και πάντοτε σημαντικό θέμα η τρομοκρατική επίθεση στην πτήση των Northwest Airlines για το Detroit επιβεβαίωσε ότι είναι πραγματική η απειλή. Θα ήθελα δε να τονίσω ότι τα υπάρχοντα πρότυπα για την ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές εφαρμόστηκαν σωστά στο αεροδρόμιο του Σίπχολ στο Άμστερνταμ. Υπήρξε όμως έλλειψη πληροφοριών και διασυνδέσεων. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός αυτό. Πρέπει επομένως στα πλαίσια της ασφαλείας να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές που την αφορούν. Όλοι οι εταιρείε, το κοινό μας ρωτούν εάν είναι επαρκή τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ή αν χρειάζονται περισσότερα οι νέες τεχνολογίες σάρωσης συζητιούνται για αυτόν τον λόγο. Οι σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια θεωρούνται από τους εμπειρογνώμονες ότι δείχνουν καλύτερα τα ύποπτα υλικά από τους υπάρχοντες σαρωτές με τις ακτίνες χ. Ποιο είναι το κόστος που αντιπροσωπεύουν όμως και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία δεν είναι ακόμη γνωστό. Το Κοινοβούλιο το 2008 είχε ήδη παρατηρήσει ότι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας αρωτών σώματος θέτει διάφορα προβλήματα εκτός από την ασφάλεια. Τον Απρίλιο θα σας υποβάλω μία έκθεση για την τεχνολογία τέτοιων σαρωτών στα αεροδρόμια για να ανταποκριθώ στο ψήφισμά σας που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσον οι ανησυχίες αυτές θα λυθούν καλύτερα σε εθνικό ή σε ενωσιακό επίπεδο. Για μένα ένα ενωσιακό πλαίσιο θα ήταν καταλληλότερο και αυτό το λέω με βάση την εμπειρία μας μιας κοινή προσέγγισης αντιμετώπιση των απειλών από την 11η Σεπτεμβρίου και, μετά. Ένα ενωσιακό πλαίσιο εγγυάται ομοιόμορφα πρότυπα και για την ασφάλεια και για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων. Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η ασφάλεια στα αεροδρόμια είναι θέμα πολύ ευρύτερο από ότι απλώς καινούργιοι σαρωτές. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην αεροπορία πρέπει να γίνει με συνδυασμένα μέτρα και καλύτερη συλλογή πληροφοριών και άλλες μεθόδους έρευνας και διεθνή συνεργασία. Όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, αφού αναπτύσσονται οι τρομοκράτες πρέπει να αναπτυχθούμε και εμείς. Αφού προοδεύουν μάλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Της Επιτροπής κυρία Μάλστρομ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Αυτό είναι η νέα διφύ προσέγγιση της Κομισιόν. Η συζήτηση έδειξε πως έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα και έχουμε ένα νέο πρόσωπο και είμαι πολύ ευτυχής και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που θα συνεργαστώ μαζί σα για θέματα ασφάλεια και για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Αυτό θα το κάνουμε σεβόμενοι βέβαια ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που έχουν τελική ευθύνη για κάθε επιχειρησιακή ε, και αντικατασκοπική εργασία σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σα θυμίσω και ορισμένοι ήσασταν στην ακρόασή μου ε, σε, πριν από κάποιε εβδομάδε, ότι στο πρώτο βήμα θα ζητήσω από τι υπηρεσίε μου να κάνουν μια αξιολόγηση για το τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Ε, ε, από αυτές τις βάσεις θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε. Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ε, ότι αυτό που έχουμε, το, το τι έχουμε, το τι λείπει και το τι επικαλύπτεται, ώστε να προτείνουμε τα νέα μέτρα πιο αποτελεσματικά. Και θα σας ε, ενημερώσω για αυτή την ε, αξιολόγηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν ε, γνωρίζω το γεγονός ότι η απειλή τρομοκρατική δεν έχει μειωθεί. Γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος κύριος Κάλλας και η Προεδρία του Συμβουλίου γνωρίζουμε πως η τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο σημαντικές αξίες για τη δημοκρατία μας. Έχουμε στατιστικές από την Ευρωπόλ που δείχνουν πως μόλις το 2008 τα κράτη-μέλη έδειξαν πως ε, Υπήρξαν τουλάχιστον 350 ε, ε, τρο, ε, τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες αναχαιτίστηκαν εντός της Ένωσης. 359 άνθρωποι συλλήφθηκαν σε σχέση με την τρομοκρατία. 50% φαίνεται πως ανήκαν στην Αλκάιντα και 39% σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η ΕΤΑ στην Ισπανία. Και ξέρουμε πως το 2008 είχαμε τα τραγικά γεγονότα και τις φοβερές ε, τη φοβερή επίθεση στο, στη Βομβάη. Ξέρουμε ότι είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μένουμε σε επιφυλακή και να μεριμνούμε ώστε να γίνονται πλήρως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να δούμε τώρα τα μέσα που έχουμε σήμερα. Έχουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη ε, τρομοκρατία. Είναι μια στρατηγική, μετά από τι ε, επιθέσει στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη, είναι μια στρατηγική ε, που στόχο έχει να καταστήσει την Ευρώπη ασφαλέστερη και να επιτρέψει στους πολίτες της να ζουν σε ένα, μια, ένα χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία άνεφας ασφαλείας και ε, φαίνεται να υπάρχει ανάγκη βέβαια για να είμαστε βέβαιοι ότι οι άλλες πολιτικές ε, θα είναι βιώσιμες και γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει μέτρα τα οποία θα εξακολουθήσουν να υπόκειται στην ε, έλεγχο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένο το αντίκτυπο στη προσωπικά στοιχεία και στους ε, ανθρώπους. Η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και γι' αυτό και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεργασία με τους ε, συμμάχους και εταίρους μας καθώς και τους διεθνούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε σχέση με την εσωτερική διάσταση της ε, αναχέτηση και της πρόληψης της τρομοκρατίας υπάρχει μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας ορισμένου στόχοι κλειδιά για το πώς θα συμβάλλουμε στην ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εγώ συμμερίζομαι απόλυτα αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει να εμποδίσουμε την ε, ριζοσπαστικοποίηση της βίας, να στηρίξουμε τα θύματα, να ανταλλάξουμε πληροφορίες ανάμεσα στις εθνικές αρχές και συνεργασία με όλους τους ε, κατάλληλους φορείς. Θα πρέπει να αντιδράσουμε στις μη συμβατικές απειλές, να βελτιώσουμε την ανείχνευση των απειλών, να στερήσουμε τους τρομοκράτες από τους οικονομικούς τους πόρους και να επενδύσουμε περισσότερη έρευνα στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτές οι εξελίξεις και αυτές τις πολιτικές φυσικά στηρίχθηκαν στεναρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου η Κομισιόν έχει κάνει μια μεγάλη συμβολή για να προσεγγιστούν τα νομικά πλαίσια των κρατών μελών ω προ αυτό. Έχουμε φτιάξει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη που θέσπισε ένα νέο δικαίωμα ε, και ορίσε, μάλλον διευκολύνει τι διαδικασίες έκδοσης ανάμεσα στα κράτη τη Ένωση. Έχουμε επίση σημαντικέ δραστηριότητε για να ανεχνεύσουμε τρομοκρατική χρήση του ίντερνετ και να εντοπίζουμε του τρομοκράτες, ξεκινώντα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία της των κρίσιμων υποδομών και περιορίζοντα την πρόσβαση των των τρομοκρατών στην, στα μέσα που χρειάζονται για να ε, φέρουν σε πέρα τις ενέργειές τους, δηλαδή τη χρηματοδότηση και τα εκρηκτικά. Επίσης θέλουμε να μπορούμε να αναχνεύσουμε καλύτερα τους τρομοκράτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά για μια επίθεση αλλά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και ώστε να μην μπορούν να κατασκευάσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ε, αυτό θα το κάνουμε το, φέτος. Είχαμε και το πρόγραμμα δράσης CBN που προτάθηκε από την Κομισιόν και συμφωνήθηκε από, την Κομισιόν, από το Συμβούλιο πέρυσι εδώ, εκεί συμπεριλαμβάνονται 30 συγκεκριμένα project και η Κομισιόν έχει προβλέψει 30 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολύνει την εφαρμογή όλων αυτών. Η δική μου δέσμευση είναι πως τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αναπτύσσει το ρόλο της ως διευκολυντής και καταλήτης για τη συνεργασία για την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, για τη συγκέντρωση των πόρων, τη βελτίωση της έρευνας και την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων για τις ε, διεθνείς αλλαγές. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας. Μπορεί αυτό να διευκολυνθεί δημιουργώντας ε, ε, ένα διεθνές ταμείο για την ασφάλεια. Είναι κάτι που προβλέπεται από το πρόγραμμα της Οκχόλμης. Σε μεγάλη κλίμακα βέβαια διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την ε, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών. Χιλιάδες χιλιάδων πολίτες ε, μπλέκονται εδώ και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και εδώ αυτό φάνηκε στην τελευταία συζήτηση που είχαμε ε, ψηλά στάνταρα προστασία των δεδομένων ε, για να μην υπάρξει κατάχρηση κακοδιαχείριση των στοιχείων. Και σα σας διαβεβαιώνω πως ε, εξετάζουμε το θέμα δεόντω και μαζί με τη συνάδελφο Ρέντινγκ θα υποβάλουμε στο εγγύ μέλλον ένα καθεστώ προστασία που θα καλύπτει και τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση και θα καλύπτονται από την ομπρέλα της στρατηγικής εσωτερική ασφάλειας την οποία θα σας υποβάλουμε σε ε, συντόμως. Και ε, τέλος, Πρόεδρε, να καταλήξω ότι μακροπρόθεσμα μπορούμε να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία αν είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε για τις αξίες μας και να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν πρέπει οι πολιτικές μας να, να γίνουν αντιληπτές ως αμφίσιμες ή ότι χρησιμοποιούν διπλά μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει να προλάβουμε την αποξένωση στις κοινωνίες στις οποίες ζητούμε αν είμαστε πιστοί στις αξίες μας, στη δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ελπιδοφόρα η προοπτική σας. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, θα έχουμε και τον κύριο Κάλλας και εσάς μαζί. Ε, θα είμαι πολύ αυστηρός με τον χρόνο, κύριε Βέμπερ. Το καταλάβατε αυτό, φαντάζομαι, στα ελληνικά, όπως το είπα. I will be very strict with the time to everyone. Ο κύριος Βέμπερ για 1,5 λεπτό τώρα ξαφνικά θα είσαστε αυστηρός με το χρόνο στους ε, ευρωβουλευτές ε, και προς την Επιτροπή, αγαπητή Επιτροπή, χαίρομαι που σήμερα δεν κάνουμε λόγο μόνο ειδικά για τους αρωτές αλλά έχουμε μια γενικότερη συζήτηση με στο οποίο συζητάμε η απειλή τη τρομοκρατία είναι πραγματική χειροπιαστή, μια απειλή για του πολίτε στην Ευρώπη. Οι δράσει που ακολουθήσαμε και υιοθετήσαμε είναι θετικέ. Και στι αρχέ μα θέλω να ευχαριστήσω τι αρχέ και τι υπηρεσίε. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για θέματα ασφάλεια έκαναν καλή δουλειά μέχρι σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσουμε γι' αυτό τώρα, να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον. Τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και εδώ τρεις συγκεκριμένες παρακλήσεις ή αιτήματα θα είχα. Πρώτον, συνεργασία των αρχών μεταξύ τους στην Ευρώπη. Σε κάθε έγγραφο αναφέρεται πηχιαία ότι πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία. Εξαιρετικές δηλώσεις όμως χειροπιαστά δεν γίνεται τίποτα. Και στο Τολέδο πάλι δεν έγινε τίποτα σε σχέση με τη χειροπιαστή πρακτική συνεργασία. Δεν απουσιάζουν δεδομένα και στοιχεία, αλλά απουσιάζει λύπη η συνεργασία των αρχών. Παρακαλώ το Συμβούλιο να κάνει τη δουλειά του και να υποβάλει και η Επιτροπή της αντίστοιχε προτάσει για να προωθηθεί αυτό. Δεύτερον, ο προβληματισμό σε σχέση με τη συλλογή στοιχείων για το κινητό τηλέφωνο, για παράδειγμα, την αποθήκευση τέτοιων στοιχείων και να αποτελέσει το νομοθετικό πλαίσιο λιδία λίθο από πλευρά του ΕΛΚ πρέπει νομοθετικά να παρακολουθήσουμε αυτέ τι εξελίξει ε, και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τρίτον, είχαμε τη συζήτηση για το SWIFT ε, μόλι πριν. Παρακαλώ να σκεφτούμε γιατί θα πρέπει να διοργανωθεί η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να διοργανωθεί με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είμαστε εμεί σε θέση ω Ευρώπη να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε αυτά τα στοιχεία. Και εδώ πάλι τίθεται το θέμα. Αυτό θα ήταν μια ιδέα για να προβληματιστούμε για το μέλλον, τι πρέπει να γίνει και ζητώ συγγνώμη αν ξεπέρασα το χρόνο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγο χρόνο μου δώσανε και εξ ονόματο της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σα πω ποια είναι τα βασικά κριτήρια και προαπαιτούμενα και για το σαρωτή σώματος που μέχρι πρόσφατα μας λέγανε ότι ήταν πανάκια και το θαυμαστό μέσο. Χρειάζεται εναρμονισμένη προσέγγιση ευρωπαϊκή, με ευρωπαϊκούς κανόνες παιχνιδιού. Αλλιώς ε, δημιουργούμε ένα χάος, ε, μετατοπίζουμε το πρόβλημα ασφαλείας και θέλω να πω στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι στο μεταξύ κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες. Δεύτερο, χρειαζόμαστε ενιαία προσέγγιση, συνολική όχι βεβαιασμένα ε, συμπεράσματα, όχι εξαγγελίες και ο ερωτήσει του σώματος να είναι ένα στοιχείο ευρύτερης πολιτικής με συνοδευτικά άλλα μέτρα και άλλα στοιχεία όπως είναι η δημόσια υγεία και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις. Και ένα τρίτο, θα πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε την εντύπωση ότι το σαρωτή σώματος είναι ε, υποτιθέται 100% ασφαλής το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βρίσκει εκρηκτικά επάνω στο σώμα. Αλλά όχι στο ιστορικό του σώματος. Ωραία. Υποστηρίζω και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει πρώτα μελέτες και μετά πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάιζνερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ο Υπουργό Πέρεθ Ρουμπαρκάμπα το είπε σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ασφαλέ σύστημα για τι εναερίε μεταφορέ. Θέλουμε να έχουμε ασφάλεια σε εναερίε μεταφορέ. Το Ντιτρόιτ και το Μίνχεν, το Μόναχο στη Γερμανία έδειξαν ότι υπάρχουν κενά. Και γι' αυτό τώρα έχουμε αυτή τη βιασύνη να χρησιμοποιηθεί το μέσο των σαρωτών σώματο. Υπάρχουν αυτοί στι ΗΠΑ και αλλού. Τώρα το ερώτημα τίθεται, θα είναι πιο ασφαλή οι εναέριες μεταφορές. Αυτό είναι το αποφασιστικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε. Στους σαρωτές σώματος υπάρχουν πολλά ζητήματα που τίθενται. Ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται, τι είδου ακτινοβολία χρησιμοποιείται, είναι βλαπτική για την υγεία, τι μπορεί κανείς να δει, κάποια κόκκινα και πράσινα σημεία ως στιγμές ή και το σώμα. Διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά κοστίζουν και χρειάζεται και χρόνος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να προσαφινιστούν. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε θέλετε εσεί να το κάνετε και να υποβάλλετε πρόταση. Χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση σχετικά. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Τελαβίβι ή καμιά άλλη μέθοδο θα, να αναζητηθεί δηλαδή ο ε, κομιστής των εκρηκτικών και όχι μόνο το εκρηκτικό, τα εκρηκτικά. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν διασφαλίζοντας τα δικαιώματα όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο εδώ και καιρό διαπιστώνει ότι αν φέρουμε τους ερωτές ε, σώματος θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές, προστασία των δεδομένων της ανθρώπινης εξοπρέπεια της ιδιωτικής σφαίρας, ελευθερία επιλογής, δημόσια υγεία. Υπάρχουν τεχνικές που τα εγγυώνται όλα αυτά πλέον, αλλά φοβούμε ε, ότι αυτές οι ε, εντυπώσεις που κυκλοφορούν είναι ότι θα υπάρχουν ε, φωτογραφίες ε, γυμνές. Αυτά χρησιμοποιούν ε, στο Λονδίνο και δεν δίνουν ελευθερία επιλογής. Στην Ιταλία έχουν νέα τεχνολογία και το Ολλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητάει να υπάρχουν σαρωτές σώματος για παντού, όχι για τις πτήσεις μόνο προς τις Ηνωμένες δεν θα πρέπει να συζητάμε τα τεχνικά θέματα. Την ουσία βοηθάει αυτό, βοηθάει την κοινωνία. Εγώ συμφωνώ αυτό που είπε ο συνάδελφος σοσιαλδημοκράτης και ε, έθεσε και τις ερωτήσεις αυτές. Θα πρέπει να δούμε τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Και η πλήρης ασφάλεια δεν υπάρχει 100%. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάλεν για λεπτό. Πρόεδρε η πιο πρόσφατη ε, γενιά σαρωτών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Έχουμε ε, ε, μόνο ένα σχεδιάγραμμα του ανθρωπίνου σώματος και μια μηδρή εικόνα αν κάποιος έχει πάνω του όπλα εκρηκτικά ή άλλα απαγορευμένα στοιχεία. Και αν τους βρούμε αυτούς τότε τους ελέγχουμε ξεχωριστά. Και επίσης δεν θίγουν και τη δημόσια υγεία είναι η ακτινοβολία τους χαμηλότερη από εκείνη των κινητών τηλεφώνων. Και επίσης ε, ε, μειώνονται και οι ε, χρόνοι αναμονής γιατί με τους αρωτές αυτούς περνάνε πιο γρήγορα οι επιβάτες. Οπότε, Πρόεδρε, αυτά τα στοιχεία όμως δεν είναι πανάκια. Και το profiling και η καλή πληροφορία είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Είναι συμπληρωματικοί μόνο οι σαρωτές. Είμαι υπέρ, αλλά να είναι συμπληρωματικά αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ταβάρας για λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μερικέ μέρε έλαβα ένα email από κάποιον ομάδα πίεση που πουλάγε σαρωτέ σώματο. Και είναι αλήθεια ότι κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα κοστίζει 250.000 ευρώ. Μια ολόκληρη περιουσία. Αλλά. Το να περνάει ο κάθε τουρίστας από εκεί μέσα και, από, και όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να δούμε αν τελικά πρόκειται, ε, αν θέλουμε μάλλον τέτοια εμπορεύματα να χρησιμοποιηθούν. Ε, δεν μπορούμε όμως να τα χρησιμοποιούμε τα πάντα για να αυξάνουμε διαρκώς τα επίπεδα παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή του καθενός. Εμείς εδώ στο Κοινοβουλίο έχουμε ευθύνη, εντάξει, να, αν είναι αλήθεια ότι η αστυνομία χρειάζεται διαρκώς περισσότερα στοιχεία, είναι σημαντικό να βασίστη η έρευνα αυτή σε βέβαιες υποθέσει υποθέσεις. Και υπάρχουν εδώ πολλές υποθέσεις από πλευρά του Συμβουλίου και από τις Κομισιόν που είναι λανθασμένες. Η ιδέα δηλαδή ότι η, η τρομοκρατική απειλή δεν μειώθηκε είναι αμφισβητήσιμη και πρέπει να τη συζητήσουμε εδώ. Η ιδέα ότι η τρομοκρατία εξελίσσεται και εμείς πρέπει και να εξελιχθούμε. Αλήθεια. Αλλά αρχίστε από το να κάνετε καλά τη δουλειά σας γιατί η, προσπά... η απόπειρα ε, στο Detroit θα μπορούσε να έχει αποφευθεί πολύ εύκολα. Δηλαδή, πρέπει να, να συζητήσουμε τις βάσεις δεδομένων του μέλλοντος. Όταν ε, ανακαλύφθηκε πως οι τρομοκράτες μπορούν ε, να καταπιούν τους, τους ε, εκρητικούς μηχανισμούς, τι θα, βάλουν τους, βάλουν τους αρωτές. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε ένα σημείο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα europos parlamentas privalo padaryti viską kad e, slaptųjų tarnybų πρέπει... να καταβάλει κάθε προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> στην ε, χρήση αυτών των μέτρων κατά της τρομοκρατίας να μην χρησιμοποιούνται ε, κρυφές ε, φυλακές ή άλλα μέτρα ε, βασανισμού και σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν από πλευράς του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου εκεί έδωσε μαρτυρία για βασανιστήρια στο Ουσμπεκιστάν. Γνώριζε για το φάκελο κάποιου που είχε συλληφθεί επειδή τον ε, έβαλαν ε, μέσα σε ε, μια δεξαμενή με βραστό νερό και επίσης ε, στοιχεία σε σχέση με, ε, που αντλούνται από, ε, μετά από βασανιστήρια χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη αντίφαση σε σχέση με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν με βασανιστήρια αντλούνται τέτοια στοιχεία. Θα ήθελα να επανασυσταθεί η προσωρινή επιτροπή σε σχέση με τις παράνομες συλλήψεις από CIS στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κ. Κλάις Προσοχή η συζήτηση κατά της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να ε, καταντήσει συζήτηση για τους αρωτές ή τα προσωπικά δεδομένα. Μας κάνει εντύπωση που το Συμβούλιο και η Επιτροπή στη δήλωσή τους δεν μίλησαν για τον ακραίο ε, Ισλαμισμό που είναι πρόσφορο έδαφος και ε, καλλιέργεια του ε, ε, νέου είδους τρομοκρατίας. Αυτή την πραγματικότητα αν δεν τη βλέπουμε τότε είναι καταδικασμένη οποιαδήποτε προσέγγιση από την αρχή να αποτύχει. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο μιλάει για τα δικαιώματα, τα πολιτικά και καλά κάνει. Αλλά χανόμαστε ε, μέσα στα τυπικά αυτά και ε, καλλιεργείται ε, μια φοβία απέναντι σε οποιαδήποτε προσέγγιση κατά της τρομοκρατίας και δεν εξυπηρετούμε έτσι τους πολίτες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους υπόλοιπους συγγραμμένους ομιλητές. Ο κύριος ε, Κούν για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι για το ΕΛΚ και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι η κυριότερη πρόκληση του 21ου αιώνα και έτσι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο στην Επιτροπή Μεταφορών όχι μόνο έχουμε και διατάξει ρυθμίσεις ε, για την απαγόρευση ε, ρευστών ε, και υγρών στις αποσκευές αλλά και εξετάζουμε και τα θέματα σαρωτών σώματος και ένα πράγμα υπονοημίου πρέπει να πω 100% ασφάλεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ούτε και στο μέλλον μπορεί να διασφαλιστεί φυσικά μπορούμε να εκπονήσουμε και να αναπτύξουμε τεχνικές και τεχνολογίες που μπορούν να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν μια μεγάλη μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά προ το 100% δεν μπορεί να είναι ποτέ πάντα απόλυτη. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι συμφωνούμε διακομματικά ότι πρώτον η υγεία των επιβατών το δυνατόν δεν πρέπει να ε, πληγεί και να υποστεί κάποιε αρνητικέ επιπτώσει. Πρέπει να αναπτυχθούν με καλή βάση τέτοιου είδου εξοπλισμοί όπω οι σαρωτέ σώματος με μια καλή πρακτική. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να διασφαλίζονται αυτέ οι πτυχέ και όχι μόνο σαρωτέ σώματο να λειτουργούν σαν παράδειγμα όπου με ακτινοβολία θα μπορεί κανείς να δρά αλλά και στην Επιτροπή Μεταφορών έχουμε και αποκοινούμε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, προβληματιστεί και συμφωνήσει και είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για τους ε, σαρωτέ σώματος κατά τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε πριν από τις ερηνές διακοπές και πρέπει να διασφαλίσουμε μια συνεκτική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών που είναι αρμόδια επί της και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για την συμβατότητα των, τεχνολογικών μέτρων και την πιστοποίηση, αδειοποίηση και παντού πάντα ήδη όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών των συσκευών ώστε να μπορέσουν πανευρωπαϊκά να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι ήταν τρεις οι επίτροποι που είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα εδώ παρόντες και χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλλά να σας πω και ποια αποσιάζει. Επίτροπος Ρέντινγκ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι σαρωτές σώματος μπορεί να ε, επηρεάσουν ενδεχομένω την ιδιωτική σφαίρα και θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε σε βάθος τον αντίκτυπό του. Τέτοια ακριβώς πράγματα δεν πρέπει να λέμε ε, στην αρχή ε, της προσπάθειας. Εμείς ως δημοκράτες πιστεύουμε ότι τα τεχνικά μέτρα βοηθούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η κυρία Μάνστρομ καλά τα είπε. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Εγώ ε, έχω πολλές φορές ε, εμποδιστεί να ταξιδεύσω σε αεροδρόμια. μου επιτρέπει η τεχνολογία να ταξιδεύω καλύτερα, ε, τόσο το καλύτερο. Και έχω και ανθρώπους από την εκλογική μου περιφέρεια που τους στιγματίζουν, που τους ελέγχουν ιδιαίτερα. Ε, χρειάζεται κοινή προσέγγιση, καλή τεχνολογία, βεβαίως και η προστασία των ελευθεριών. να μην υπάρχει κανένας αδύναμος κρίκος σε κανένα αεροδρόμιο. Τα κράτη-μέλη που το ξεκίνησαν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πανευρωπαϊκή προσπάθεια και ασφαλή. Η κυρία Λάτφορντ για ένα λεπτό. Oh, ναι. Αρχίζω ξανά. Θέλω να μιλήσω για το κράτος δικαίου και οι μυστικές υπηρεσίες που δεν τα σέβονται αυτά. Ε, έδειξε μια σημερινή δικαστική απόφαση στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο ε, ότι οι μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν και ε, συνεργάστηκαν στην υπόθεση του Μπενιάν Χαμίτ που είχε κρατηθεί σε μυστική φυλακή και είχε κακοποιηθεί. Πού είναι ε, η συνθήκη κατά των βασανιστήριων. Το 2006 ε, εγώ ήμουν επικεφαλής σε μια επίσκεψη στο Λονδίνο της αντίστοιχης επιτροπής. Ο τότε υπουργός Τζεφ Χούν Στη μισή συνεδρίαση ε, μου απαντούσε επιμόνως ότι κάνουμε έρευνες για το κατά πόσο υπήρχε ε, συμμετοχή ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Μου είπες πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη κάποια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο πλήρης ανεξάρτητη έρευνα χρειάζεται ε, για το κατά πόσο συνεργάστηκε η κυβέρνηση ε, ε, του εργατικού κόμματος σκυλάκι του Μπούς στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δούμε, να αποκαλυφθεί τι εντολές δόθηκαν στους πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου για να σιωπούν σε περιπτώσει βασανιστήριων και πλήρης κοινοβουλευτικό έλεγχος που δεν τον έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις μυστικές υπηρεσίες. Ο κύριος Μπράντμπερν για ένα λεπτό. Uh, um, Ευχαριστώ. Να επανέλθω στους αρρωτές σώματος. Οποιοδήποτε μέτρο που αυξάνει την ασφάλεια του κοινού που ταξιδεύει είναι καλοδεχούμενο. Πριν όμως θα πρέπει να είναι και ε, ανάλογη η προσέγγιση, όχι δυσανάλογη. Και να ε, έχουν και το σεβασμό που τους ανήκει οι ε, επιβάτες. Είδαμε τα Χριστούγεννα την απόπειρα αυτή την τρομοκρατική που ευτυχώ να βάγει. Θα πρέπει να αυξηθεί η ασφάλεια με οποιοδήποτε τρόπο και σε κάποια κρατημέλη, ειδικά ε, στο δικό μου, η χρήση ε, τέτοιων ε, μηχανημάτων είναι τώρα υποχρεωτική. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. No scan, no fly. Δεν σαρώνεις, δεν πετάς. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει σκανδαλώδη τακτική, δεν προστατεύονται καν τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις τα Χριστούγεννα είδαμε ότι ξανά άνοιξε ε, αυτό και είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι δεν ήταν ζήτημα ασφαλείας στο αεροδρόμιο αλλά ήταν ζήτημα κακής συνεννόησης των μυστικών υπηρεσιών που δεν αντέλεξαν τις πληροφορίες που έπρεπε. Και δυστυχώς πρόεδρε πρέπει να πω τελειώνοντας ότι τώρα θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα profiling των επιβατών. Κύριος Μπορκέζιο, για ένα λεπτό. Il terrorismo evolve τρομοκρατία, βόμβες, εμείς πρέπει να τρέχουμε από πίσω, από πίσω από τις ε, σχηματισμούς τους τρομοκρατικούς ε, που είναι δύσκολο να ανοιχνεύσουμε. Και εμείς εδώ μιλάμε για ιδιωτική ζωή, για το αν θα πρέπει να υιοθετήσουμε πιο προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους. Αντίθετα θα έπρεπε να ανησυχούμε για ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, το οποίο νόμα αποφασίζει αντί να, αντί να αποφασίζει για να βοηθήσει, να αποφασίζει να, αποδυναμ, να μας αποδυναμώσει απέναντι στην τρομοκρατία, την Ισλαμική τρομοκρατία. θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί υπάρχει όλο ένα και πιο μεγάλη απειλή. Τη στιγμή που οι τρομοκράτες τόσο δύσκολο είναι να ανέχνευθούν και να αντιμετωπιστούν, τι body scanner και σαχλαμάρες, εδώ μπαίνουν παντού. Μπορεί αύριο το πρωί να μπουν στο αεροπλάνο που εμείς θα πάρουμε. Αν ε, εμεί ε, υποχωρήσουμε με τις υπερβολικές εγγυήσεις, ε, ανοίξουμε ένα μεγάλο κενό για την εσωτερική ασφάλεια των χωρών μας και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε με την Επίτροπο. Δεν πρέπει να είμαστε να γενικεύουμε με αυτόν τον κακό ε, Ισλαμικό τρομοκρατισμό. Ευχαριστώ πολύ. Το 2000 2.000 άνθρωποι παγκόσμια λόγω τέτοιων τρομοκρατικών αποπειρών απεβίωσαν. Σε λίγα χρόνια 16.000 και στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε 6.000 ανθρώπους που καθημερινά αποβιώνουν λόγω AIDS. Πρώτον, η τρομοκρατία είναι μια ιστερία που οδηγεί στο να χρησιμοποιούνται για παράδειγμα τώρα σαρωτές σώματος. Αυτού του είδους η καταπολέμηση τη τρομοκρατίας απέτυχε. Το πρόβλημα το ενέτεινε ακόμα παραπέρα. Όσον αφορά τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να πω ότι αυτή η Ευρωβουλή κατεπηγόντω θα πρέπει να ασκήσει δικαιώματα κοινοβουλευτικού ελέγχου όπως σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης θέλω να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισαγωγή των κοινών προδιαγραφών για το user interface. Εδώ θα πρέπει να προαχθεί αυτή η συνιστόσα. Η χρηματοδότηση πρέπει να διασφαλιστεί γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Χιμένες για ένα λεπτό. Ναι, πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σε ένα θέμα τόσο σοβαρό σαν την τρομοκρατία δεν θα πρέπει να αναμένουμε τα γεγονότα για να δράσουμε. Θα πρέπει να τα προλαβαίνουμε και να δούμε πιο πριν. Να δεν το κάνουμε. Και δυστυχώ, όπω αυτή την απόπειρα που είδαμε που απέτυχε μεν στον Τιτρόιτα, αλλά μα υποχρεώνει να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στι εναερίες μεταφορές. Η χρήση σαρωτό σώματο στα αεροδρόμια είναι μια ευθύνη που δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε. κυρίε και κύριοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε, διότι δεν περιμένουν, δεν αναμένουν οι τρομοκράτε. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου και δεν θα υπάρχουν ε, βλαπτικές επιπτώσει για την υγεία. Θα πρέπει να ληφθούν πανευρωπαϊκά οι, αρμο... οι ε, αποφάσεις. Ε, για, την περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πω δεν υπάρχει κανένα ανώτερο δικαίωμα από το δικαίωμα στη ζωή και το, όταν θέτουμε την ελευθερία πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Λόπεζ Αγγιάρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η τρομοκρατία είναι μια παγκόσμια απειλή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού όλοι. Είναι ευθύνη μα. Γι' αυτό η συνθήκη τη Λισαβόνα, που είναι η βάση για να διασφαλίσουμε μια κοινή πολιτική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία στην Ευρώπη, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη συνένεση. Από ό,τι άκουσα από την Προεδρία του Συμβουλίου κάποιες από τις συνιστώσεις ε, που πρέπει να είναι στη βάση αυτής της κοινή πολιτικής είναι πρώτον η ενίσχυση της ε, κοινή πληροφόρησης και ενημέρωσης ε, για να αποφύγουμε τέτοιου είδους απόπειρες και να ανοιχνεύουμε τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Δεύτερον, να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε όλες τις τεχνολογικές προόδους και μέσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ανάλογη σχέση με την διασφάλιση των προσωπικών δικαιωμάτων των πολιτών. Μετά, σε σχέση με κάποιες χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το κέρας της Αφρικής ε, να δούμε ειδικά την αντιμετώπιση της τρομοκρατία. Η τεχνολογική πρόοδος των, των σαρωτών σώματος θα πρέπει να είναι συμβατή με την ανθρώπινη υγεία, αλλά να μην αποβαίνουν ποτέ όσον αφορά τα αεροδρόμια, να μην είναι ποτέ ει βάρο ε, των επιβατών. Πρώτον, πρέπει να δούμε το κόσι, την Επιτροπή. Δεύτερον, ε, σε σχέση με το Συμβούλιο που έγινε στο Τολέδο και το διατλαντικό χώρο ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει μια πολύ ασφαλή συνεργασία με τις ΗΠΑ μέσα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των κοινών απειλών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ένας από τα μέσα πρόληψη της τρομοκρατίας είναι η πληροφορία. Θα πρέπει όμως να κυκλοφορεί η πληροφορία αυτή. Συμβαίνει αυτό σήμερα. Τίποτα δεν είναι λιγότερο σίγουρο. Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ενημερώνουν του Ευρωπαίους Ομολόγου τους. Πάντως για το ε, φερόμενο τρομοκράτη που ε, συνελήφθη στη πτήση Άμστερνταμ-Διτρόιτ χωράνε αμφιβολίες εδώ. Και γενικά θα πρέπει να αναρωτηθούμε με αφορμή αυτό εάν το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών στη δρομοκρατία σέβεται την αρχή τη αμοιβαιότητα. Ένα όργανο κοινοβουλευτικού ελέγχου επιβάλλεται ε, επιγόντω. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε από το κοινοβούλιο μας να ε, δίνει όλο και περισσότερο ε, προσωπικά δεδομένα η Ευρώπη, αν ε, αντίστροφα οι αμερικανικές αρχές δεν δίνουν ουσιαστικές πληροφορίες στις δικές μας υπηρεσίες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό χρειάζεται και επιβάλλει μια επιτροπή κοινοβουλευτική ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιζότο για ένα λεπτό. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μιλάμε για καταπολέμηση τη τρομοκρατίας συζητώντα μόνο για ε, κατασκοπία και τεχνολογία έχω την εντύπωση πω ε, εξετάζουμε το θέμα με κατάλληλο τρόπο. Λε και θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε μια αρρώστια επικεντρώμενη επικεντρωνόμενοι μόνο στα συμπτώματα ε, και όχι στα αίτια σας. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε στην καρδιά του θέματος, όχι μόνο στην εξωτερική της ε, εικόνα. Το να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα θα, σημαίνει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την τρομοκρατία που είναι άμεση εκδήλωση της ανικανότητας ή της, ε, της μη βούλησης από πλευρά των εθνοτικών ομάδων να ενσωματωθούν στον ευρωπαϊκό ιστό. Εγώ διερωτώ με λοιπόν και ρωτώ το Κοινοβούλιο, θέλουμε να συζητήσουμε για την τρομοκρατία, έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε πολιτικά μια συζήτηση για την ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη και για το αν συμμερίζονται αξίες και ε, δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε με, για το ηθικό σκέλος του θέματος. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει βούληση για τη μετώπιση του θέματος. Σας ρωτώ συνάδελφοι όλων των πολιτικών ομάδων, αν όχι σε αυτό το θέμα, σε ποιο άλλο θα πρέπει να δείξουμε συνεργασία και πολιτική ε, βούληση. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος της Βόρειας Ιρλανδίας γνωρίζω πολύ καλά τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στους αθώους πολίτες. Καταστροφή και δολοφονία στη ζωή απλών ανθρώπων που πηγαίνουν να ψωνίσουν ένα Σάββατο που, σε κλίμακα που να θυμίζει καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ μιλάμε για συνεργασία των σωμάτων ασφαλείας. Από την εμπειρία της Βόρειας Ιρλανδίας βλέπουμε ότι μπορούν να αποφευχθούν οι απώλειες ζωών από τη συνεργασία των σωμάτων αυτών και από, την καλύτερη, από τον καλύτερο συντονισμό τους. Όσοι έχουν επιλέξει την ασφάλεια έναντι της, ε, των ατομικών ευθεριών πρέπει να το ξανασκεφτούν γιατί η τρομοκρατία πράγματι καταστρέφει ζωές και άκουσα εδώ μέσα ότι η τρομοκρατία δεν είναι παρά απλή ιστερία. Αυτά είναι ανοησίες. Πιστέψτε με, όταν προσπαθεί κάποιος οπλισμένος να σας σκοτώσει δεν είναι καθόλου ιστερία το πρόβλημα αυτό, αλλά κάτι το πραγματικό. Ευχαριστώ. Είναι αναγκαίο να προστατεύσουμε ζωές και αγαθά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στα μέσα μεταφορών. Υπάρχουν εδώ ανησυχίες όσον αφορά του άρτε σώματος. Τρία από αυτά τα θέματα πρέπει να επιληθούν. Η μελέτη που ε, θα συνταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα υποβληθεί στην Ευρωβουλή. Πρώτον, είναι αναγκαίο και είναι αποτελεσματικά αυτά τα εργαλεία βλάπτουν την υγεία ή όχι παραβιάζουν τρίτον ε, την ιδιωτική ζωή ε, των ε, προσώπων έχουμε αυτές τις ανησυχίες πρώτον έλεγε, αναφερόταν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιείται είτε αυτό το σύστημα των σκάνες των σαρωτών είτε η προσωπική ε, έρευνα, σωματική έρευνα. Αλλά φαίνεται ότι καταλήγουμε τώρα στο no check no fly. Υποχρεωτική λοιπόν χρήση και όχι εθελοντική χρήση των σαρωτών. Και για την ε, χρήση αυτή θα πρέπει να ε, αναφερθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε την ευθύνη να βρούμε λύσεις που θα ενισχύουν την ασφάλεια χωρίς να διακυβεύουν την αξιοπρέπεια ή τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλοι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη δρομοκρατία και την απειλή που συνιστά κατά των δημοκρατιών μας. Αυτό είναι νομίζω συνένεση πάγια και στο Κοινοβούλιο. Μία ρίση λέει ότι ένας λαός που είναι πρόθυμος να θυσιάσει λίγη ελευθερία για λίγη ασφάλεια τελικά χάνει και τα δύο. Αυτό είναι υπερβολικό. Πρέπει να βρεθεί κάποια ε, ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, γιατί αυτό είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, γιατί αλλιώς θα έχουν κερδίσει οι τρομοκράτες, αν καταφέρουν να μας τρομοκρατήσουν όλους. Δύο ζητήματα τώρα και ερωτηματικά για το σαρωτή σώματος, για την ασφάλεια. Επιτρέπουν σήμερα οι σαρωτές αυτή αυθεντικά να έχουμε ασφάλεια και από πλευράς ε, ε, ελευθερίας, γιατί είμαι και μέλος στην Επιτροπή Ελευθεριών, διαρωτώ με πραγματικά και προβληματίζομαι αν υπάρχει πρόβλημα ε, υγείας, βεβαίως προσβολής της ιδιωτικής σφαίρας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τι γίνεται με τη χρήση των εικόνων αυτών. Ας περιμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από κοινού να προχωρήσουμε για την ασφάλειά μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Δεν θα δεχτώ λυπούμε μπλε κάρτες και θα είμαι και πάρα πολύ αυστηρό δυστυχώς στο Catch διότι δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Μπάτεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τρομοκρατία είναι χρήση βίας και εκφοβισμού για πολιτικούς στόχους. Εμείς που είμαστε υπέρ της ελευθερίας της δημοκρατίας θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε για τη τρομοκρατία γιατί πιάνει. Το Συμφέιν και ο Ήρα τώρα είναι στην κυβέρνηση στη Βόρεια Ιρλανδία. Και έβαλαν βόμβες και, και άνοιξαν το δρόμο τους μέχρι τις κάλπες με βόμβες, με δολοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες πιο άλλο, πιο εύγλωτο παράδειγμα από την τρομοκρατία, την κρατική στην Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και Σοβιετική Ένωση. Συνεχίζει η Κίνα μετά από 61 χρόνια την τρομοκρατία του Κομμουνιστικού Κόμματο. Υπάρχει καλύτερο και πιο επιτυχημένο παράδειγμα τρομοκρατία. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε και συμμετέχουν ε, και πρώην στελέχη ε, και συνοδοιπόροι και κομμουνιστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην μαοϊστές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψηφίζαμε χτες, ε, τέτοια πρόσωπα είναι. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Grazie Presidente. La sicurezza delle nostre società è un valore non negoziabile che dobbiamo perseguire con determinazione. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι διαπραγματεύσιμε οι αξίε τη Ευρώπη και πρέπει να τι διατηρήσουμε με πιο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή μάλλον η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα πρέπει να συνοδεύεται από μεγαλύτερη συνεργασία των συστημάτων πληροφόρησης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί καλώς έπραξαν που δεν παρασύρθηκαν από συγκινησιακά επιχειρήματα αλλά αποφάσισαν πρώτα να πειραματιστούν για να δουν πώς ακριβώς λειτουργούν αυτοί οι καινούργιοι σαρωτές. Πρέπει να γνωρίσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών τους όσο το δυνατόν συντομότερα, αν υπάρχουν επιπτώσεις επί της υγείας ας πούμε. Εδώ πρέπει να ισχύσει η αρχή της φρόνησης. Η έκθεση σε ακτίνες Χ είναι κάτι πιο σημαντικό από το αν είναι θέμα η σωματική έρευνα, αν δημιουργεί αισθήματα ντροπή στον ερευνούμενο. Πρέπει να κάνουμε θυσίες μπροστά στην απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας εφόσον απειλεί τη σωματική ακαιρεότητα. Αγαπητοί συναδελφοί, πια ορίστε τα ονόματα των επομένων ομιλητών. Θα τους ανοίγω το μικρόφωνο μετά από ένα λεπτό, δεν θα βαράω το σφυράκι και δεν θέλω να με παρεξηγείτε. Με τη σειρά που τους έχω. Mr. Matulka, Mr. Lightfried, Mr. Ensik, Ms. Benova, Mr. Tannock, Mr. Ernst, and Mr. Molzer. One minute each, and that's it. Apologies. Ένα λεπτό καθένας και μετά θα κλείνω το μικρόφωνο. Σαζάτα. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπό το φως της σημερινής συζήτησης, Φαίνεται ότι η εφαρμογή των σωματικών σαρωτών αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα. Το θέμα της ασφάλειας των ταξιδιωτών βρίσκεται πάνω-πάνω σε πρώτη θέση. Αλλά δεν επιτρέπει να ξεχνάμε ότι η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να τηρείται. Η εφαρμογή, η χρήση τέτοιων ε, μηχανισμών και εξοπλισμών αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ποια επιρροή ασκούν στην υγεία αυτού του είδους οι σαρωτές. Με ποιο τρόπο μπορεί η εικόνα του ατόμου που σαρώνεται από αυτούς τους σαρωτές ε, να παραμένει μέσα σε ιδιωτικά πλαίσια και να μην δημοσιεύεται. Είναι, έχει νόημα να δαπανούμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμό όταν γνωρίζουμε ότι δεν είναι σε θέση να ανοιχνεύουν εκρηκτικά. Εφόσον δεν υπάρχουν απαντήσει επαρκή, δεν επιτρέπεται εμεί να είμαστε υπέρ τη υποχρεωτική εισαγωγή και χρήση των σαρωτών. Και κάτι άλλο ακόμα επίση. Πιστεύω ότι βρήκαμε μια λύση και τώρα αναζητούμε το πρόβλημα για αυτή τη λύση που υποτίθεται ότι βρέθηκε. Αυτή η λύση λοιπόν είναι η σκάνερ. Κύριος Γιακολίνο, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω βασικά ότι το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το σοβαρό αν δεν το διασφαλίζουμε είναι πολύ ε, άσχημα τα πράγματα. Η περασμένη εβδομάδα ε, ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για το πρόγραμμα της Στοχόλμης που ζητάει εξισορρόπηση ε, μεταξύ καταπολέμησης της τρομοκρατίας και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Αν σήμερα, αν λέγω σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτά τα θέματα, τότε τότε λέγω το πρόβλημα της προστασίας τίθεται εκ νέου. Ερωτώ λοιπόν την Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάτι πρέπει να αποσαφινιστεί εκ προημίου. Μέσω αυτής της συζήτησης δεν καταδεικνύεται μόνο το ότι υφίσταται κίνδυνος λόγω της τρομοκρατίας, αλλά καταδεικνύεται ότι είναι επίση αναγκαίο να κάνουμε ένα βήμα, να είμαστε ένα βήμα μπρο από του τρομοκράτε. Η συζήτηση για την εισαγωγή σαρωτών σώματο σε όλα τα αεροδρόμια τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμω πολύ μεγαλύτερε επιπτώσει και διαστάσει. Αυτό το μέτρο είναι αντιφατικό, διότι, για παράδειγμα, σκόνες οι ουσίες που έχουν καταποθεί από τον ταξιδιώτη δεν μπορούν να ανοιχνευθούν από τους αρωτές. Ταυτόχρονα προσπαθούμε την ασφάλεια και κυρίως και την υγεία των ταξιδιωτών να την διασφαλίσουμε μέσα από αυτά τα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν ε, το, ε, τα δικαιώματα να διασφαλιστούν όσον αφορά τους ε, πολίτες μας εφόσον δίνονται εικόνες γυμνού σώματος ε, σε τρίτους. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ αυτών. Λάιχτφριντ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν πρόκειται για τις εναερίες μεταφορές και την ασφάλεια σε εναερίες μεταφορές, τότε όλο και μεγαλύτερες είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι επιθυμούν, κατοδοκούν. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους σώματος έχουμε την αρχή του ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Και γι' αυτό είτε θα υπάρξουν ευρωπαϊκέ ρυθμίσει για του σαρωτέ σώματο, ή δεν θα υπάρξουν τέτοιε ευρωπαϊκέ ρυθμίσει και δεν θα χρησιμοποιούνται οι σαρωτέ. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε την αρχή καθένα κάνει ό,τι θέλει και ο καθένα θα επιτρέπεται να κάνει ό,τι επιθυμεί. Αν όμω κάτι τέτοιο θα πρέπει να εισαχθεί, όπω οι σαρωτέ, θα πρέπει να συζητήσουμε ποιο θα το χρηματοδοτήσει και πώ. Για αυτού του κοστίζουν τεράστια ποσά και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ότι ε, ως εισηγητής για αυτό το θέμα αν υπάρξει να κινητοποιηθεί το θέμα στο Συμβούλιο διότι καταρχήν πρέπει να πούμε η δημόσια ασφάλεια είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει δημόσια να χρηματοδοτείται. Ευχαριστώ. Ο κύριος είναι εδώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου στις δευτερογενείς επιπτώσεις ε, που μπορούν να υπάρξουν και να προκληθούν από την χρήση των σαρωτών σώματος. Όταν έχουμε τέτοιου είδους ε, ακτινοβολία όπως ε, με ακτίνες Χ στις οποίες εκτίθενται οι ταξιδιώτες, οι γιατροί γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να υφίσταται τέτοια ακτινοβολία σε τακτά διαστήματα ένας άνθρωπος. Όμως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτοί οι σκάνερ, οι σαρωτές μπορούν να δίνουν μια τρισδιάστατη εικόνα του ανθρώπινου σώματος. Όμως με μεγάλο κίνδυνο για την υγεία και το σώμα των ανθρώπων που ακτινοβολούνται με αυτόν τον τρόπο. Με τον χρόνο, με την πάροδο του χρόνου μπορούν να υπάρξουν γενετικές ε, αλλοιώσεις ε, και ε, κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτιθέμεθα όταν σε τακτά διαστήματα υφιστάμεθα τέτοιου είδους ακτινοβολία δεν θα δικαιολογούσαν τη χρήση τέτοιων ε, μηχανών. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Η τρομοκρατία δεν γνωρίζει αξίες και δεν έχει ε, και άλλο στόχο παρά να θανατώνει τον πληθυσμό, να θανατώνει τον κόσμο, την κοινωνία των πολιτών και όσο γίνεται πιο φτηνά. Γι' αυτό και έχουμε τόσες αυτοκτονίες. Και είναι ε, λυπηρό που δεν μπορούμε ε, να λάβουμε μέτρα που να προστατεύουν ε, τον πληθυσμό χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματά τους και οι ελευθερίες τους. Καλό θα ήταν λοιπόν, σε περίπτωση που εγκριθούν αυτοί οι σαρωτές σώματος κάποια στιγμή, καλό θα ήταν λέγω να συζητούμε και για νομοθεσία που να ε, προστατεύει και να εναρμονίζει την προστασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καταναγκαστική ε, χρήση σαρωτών ε, στα Βρετανικά αεροδρόμια ανακοίνωσε ο Γκόρντον Μπράουν, ο Πρωθυπουργό. Είναι τρομερό πράγμα αυτό, σκάνδαλο. Και οι γυναίκε, έγκυε και παιδιά ε, περνούν από ακτίνε χ για μη ιατρικού σκοπού υγιεί επιβάτες. Είναι πάρα πολύ ε, επικίνδυνη αυτή η ακτινοβολία και μετά υφίστανται και κοσμική ακτινοβολία όταν πεθάνε. Οι μαλακοί του, στόμα, του σώματος συγγνώμη, υποφέρουν. Και ε, στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε και προσβολή του DNA και ε, ως γιατρός που ταξιδεύω και συχνά καταγγέλω αυτό το μέτρο. Και είναι και αποτελεσματικό και ευλαβερό και ελπίζω αυτά τα καταναγκαστικά η Ευρώπη να τα απορρίψει. Προφάιλινγκ των επιβατών χρειάζεται. Η κυρία Έρνστ για ένα λεπτό και μετά θα δώσω το λόγο από τους Πρασίνους στην κυρία Ριβάση. Κυρία Έρνστ για ένα λεπτό. Jetzt, jetzt Ähm, Οι σαρωτέ σώματο είναι απόλυτα σαφέ και δεν αμφισβητείται από κανένα. Είναι παρέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα. Και πρέπει εδώ να θέσουμε δύο ερωτήματα. Το πρώτο, κατά πόσον είναι αναλογική η χρήση και κατά πόσον εξυπηρετεί τον στόχο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα σαφείς απαντήσεις σε αυτό. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτό το οποίο είπε η κυρία Μάμστρομ για μια αξιολόγηση, μια αποτίμηση όλων των μέσων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτά να τεθούν στο τραπέζι προτού κάνουμε κάτι και να μελετήσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεύτερον, η κίνδυνη για την υγεία. Όλοι όσοι είμαστε εδώ θα πρέπει, ουσιαστικά πρέπει κάθε εβδομάδα επανειλημμένα να περνάμε μέσα από τέτοιου άρωτε σώματο. Κάθε εβδομάδα δύο φορέ θα πρέπει να περνάω από τέτοιου άρωτε εγώ. Είναι σημαντικό λοιπόν και θέλω να γνωρίζω κατά πόσο βλάπτει την υγεία μου κάτι τέτοιο. Και ακόμα επ' αυτού δεν υπάρχουν αποτιμήσει και αξιολογήσει. Και θα ήθελα να πω, δεν είμαι διατεθειμένη να περνάω από τέτοιου άρωτε εφόσον δεν υπάρχουν σαφεί απαντήσει. Ευχαριστώ. Είστε εδώ. Uh, Κυρία Ριβαζή, θέλετε να πάρετε το λόγο Νέου. Ναι, Ένα λεπτό έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια σύνδεση εδώ μεταξύ του σαρωτού σώματος τρομοκρατίας και της υγείας. Όταν δούμε τι κάνει η Επιτροπή για την Ασφάλεια από την Ακτινοβολία, όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου συμμετέχει η Διεθνής Υπηρεσία ε, Ατομικής Ενέργειας, όπου συμμετέχει ε, ε, και άλλος φορέας για την πυρηνική ενέργεια τι λένε ότι οι έγκυες και τα παιδιά δεν πρέπει να υφίστανται αυτό το σαρωτή σώματος ακόμα και αν οι δόσεις είναι απειροελάχιστες. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συχνότητα ε, την οποία εκτίθενται ε, οι επιβάτες, ακόμα και αν είναι μικρή, αν είναι πολύ συχνή, ε, μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνους και δυσπλασίες. Η ίδια λοιπόν δικαιολογία χρειάζεται πραγματικά να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Διεθνή τρομοκρατία επανειλημμένα μέσω παραπλάνησης ή μέσω λανθασμένων αποφάσεων μπορεί να δρά. Αν τώρα τα διάφορα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, είχαν νόημα ή όχι, δεν το εξετάσαμε. Ανταυτού, μετά από κάθε απόπειρα είχαμε περαιτέρω περιορισμού των ε, ε, ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Τώρα έχουμε και χρηματική ε, επιβάρυνση και έναντι των ΗΠΑ περιορισμοί. Όλα αυτά συμβαίνουν σε σχέση με στοιχεία και δεδομένα και εδώ οι μυστικές υπηρεσίες σε σχέση με το Αφγανιστάν για παράδειγμα και το Ιράκ. Η χρήση, η συμβατότητα και ή όχι αυτών των μέσων σε σχέση με τις προσωπικές ελευθερίες δεν απασχολεί κανένα σε σχέση με τους σαρωτές σώματος για την καταπολέμηση της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Η Ισλαμική τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί αλλά πρέπει πρέπει να τερματιστεί πια ο περιορισμός των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρώπης. Λόγος στο Συμβούλιο, στον κύριο Πέρες ε, Ρουμπαλζάμπα για πέντε λεπτά παρακαλώ ή δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Αλλά άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις όλων των ομάδων και των Ευρωβουλευτών για αυτό το θέμα. Ήταν μια συνολική, ας το πω έτσι, τοποθέτηση ε, παρεμβάσεων πάρα πολύ ε, με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαριστώ για αυτό. Θα ήθελα να τονίσω όπως έκανα και στην πρώτη μου παρέμβαση ότι δεν είμαι καθόλου υπέρμαχος εγώ του να γίνονται συζητήσεις για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο και περίπλοκο και ευαίσθητο όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μετά από τις απόπειρες ή τις προσπάθειες για μια τρομοκρατική απόπειρα. Πρέπει να εξετάσουμε, να αναλύσουμε αυτές τις απόπειρες για να δούμε τι απέτυχε σε σχέση με τα συστήματα ασφαλεία μας. Αλλά επίση ε, πρέπει να δούμε όπω επισημάθηκε ε, απόψε εδώ ότι μια σόφρον συνετή πολιτική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία πρέπει να εκπονηθεί που θα έχει μελετηθεί σωστά και που θα εφαρμόζεται με αναλογικό αποτελεσματικό τρόπο. Να μην υιοθετούμε μέτρα τα οποία θα υπονομεύουν τι αρχέ μα, διότι τότε θα κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και τονίζω πρέπει να αναλύσουμε για παράδειγμα τι έγινε στον Detroit για να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδου σφάλματα στο μέλλον. Αλλά δεν πρέπει στικτοδός βιαστικά να δράσουμε μετά από κάθε απόπειρα. Γιατί αυτό πιθανότατα θα μας, οδηγήσει, θα μας οδηγούσε στο να υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία δεν θα είχαν νόημα. Τώρα, δεύτερο θέμα. Η Ευρώπη έχει μια στρατηγική στην πολιτική καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Έχουμε μια καλή στρατηγική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια στρατηγική που αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια αποτελεσματική. Και δεν χρειάζεται παρά να δούμε μόνο τι διαφορετικέ δράσει των δυνάμεων ασφαλεία στι διάφορε χώρε μα και να δούμε μέχρι ποιου σημείου αυτέ οι δράσει πρωτοβουλίε απορρέουν από εφαρμογή αυτή τη κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία που υιοθετήσαμε πριν από κάμποσα χρόνια. Έχουμε το συντονιστή για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία που οι λόγοι του και οι παρεμβάσει του είναι πολύ ενδιαφέροντε και ενδιαφέρουσε και Συνιστώ την τελευταία παρέμβασή του στο σώμα να τη μελετήσετε προσεκτικά, γιατί καταδεικνύει μέχρι ποιο σημείο έχουμε μια στρατηγική. Μια στρατηγική που κατά τον τελευταίο καιρό προσπαθούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε και να εξειδικεύσουμε στην πρόληψη μια και στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής αυτής της πολιτικής είχαμε επικεντρωθεί στην καταδίωξη, στη δίωξη. Είναι σημαντικό να προβλέπουμε και να αποφεύγουμε απόπειρε και τρομοκρατικές πράξεις και γι' αυτό επικεντρώνουμε στην πρόληψη της προσπάθειας μας. Και το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης που ανέφερα στην παρέμβασή μου πιο πριν είναι σημαντικό να αναλύσουμε το σύνολο των πολιτικών που κάθε μια από τις χώρες μας ακολουθούν για να αποφευθεί αυτή η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων που βρίσκεται σίγουρα στη ρίζα πολλών από, αυτών, από αυτές τις προσπάθειες των τρομοκρατικών αποπειρών. Καθώς επίσης και το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών και επισημάθηκε επανειλημμένα πόσο σημαντικό είναι να μην διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία συλλήβδιν αλλά τα συγκεκριμένα σημαντικά στοιχεία για εκείνον τα χρειάζεται. Αυτού του είδους ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να με χιονοστιβάδες πληροφοριών να συντρίβουμε ένα τον άλλον, να συνθλίβουμε ένα τον άλλον. Πρέπει να γίνεται αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και βελτιωνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα. Έχουμε υιοθετήσει μια στρατηγική που η δρομολόγησή τη θα μα επιτρέψει, για παράδειγμα, τα συστήματά μα ανταλλαγή πληροφοριών να λειτουργούν καλύτερα. Και όταν κάνω λόγο για ανταλλαγή πληροφοριών, έχω υπόψη την Ευρωπόλ, την Eurojust, έχω υπόψη την λειτουργία του ΣΚΟΖΑΚ που ε, έχει αναφερθεί στην Ευρωβουλή και έχω υπόψη εν τέλει και την ανταλλαγή πληροφοριών που πρέπει να γίνεται κάθε φορά και όλο και πιο αποτελεσματική. Και τέλος τέλος αληθεύει ότι το θέμα των body scanners αρωτών σώματος είναι επίμαχο και το εξετάζουμε. Και όπως είπα στην πρώτη μου παρέμβαση και όπως είπε και η Επίτροπος πιο πριν, Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε σωστά. Και το ιδανικό θα ήταν να βρίσκαμε μια ευρωπαϊκή κοινή διατύπωση που θα ίσχυε για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά κάθε χώρα θα μπορεί να ακολουθήσει τι δικέ της πολιτικέ και διατάξει και θα είχαμε κάποιες χώρες που μέσα στο ίδιο το δικό τους ε, πλαίσιο θα μπορούσαν να ακολουθούν τις ξεχωριστές πολιτικές τους. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια κοινή θέση για αυτό το θέμα από πλευράς της Ευρώπης θα βοηθούσε πολύ. Και σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερα πιο πριν στην ας το πω έτσι, αντανάκλαση αυτής της συζήτησης είναι σημαντικό να γίνει μια νυφάλια συνετή συζήτηση με τρία στοιχεία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, η αποτελεσματικότητα αυτών των σκάνε, των σαρωτών. Είναι ή δεν είναι αποτελεσματική είναι τα όρια του. Αξίζουν ή όχι για αυτό το σκοπό που θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, είναι συμβατά ή όχι με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι πολιτικέ ελευθερίε, ατομικέ ελευθερίε των ατόμων. Είναι συμβατέ ή όχι αυτέ οι συσκευέ με την ανθρώπινη υγεία και την προστασία τη. Αυτά τα θέματα, τα τρία θέματα πρέπει να μελετηθούν. Και όταν θα έχουμε τι εκθέσει για αυτά τα θέματα στο τραπέζι, θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση όπω είναι αναγκαίο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τι παρεμβάσει που έγιναν στην Ολομέλεια. <clears throat> και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμες για τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Κάλλας έχει το λόγο. Is this, uh, is this a point of order, Ms. Ladford? Διαδικαστικό είναι κυρία Λάτφορντ. Ε, ε φροντίστε να είναι διαδικαστικό. Συγγνώμη, έθεσα άμεσα ερώτηση προς, το Συμβούλιο και θέλω απάντηση. Ε, το άρθρο 6, κατάφορη παραβίαση αυτής της διάταξης ε, της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα δεν είναι διαδικαστικό, διακόπτει ο Πρόεδρος. Μα κυρία Λάτφορντ λέει ότι είχαμε και απόφαση από το ΟΔΕ. Σάρα, ζητώ, συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Κάλλας. Ladies Um, <laughs> Αξιότιμοι βουλευτές, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας, αλλά σήμερα δεν έχουμε πρόταση για να υποχρεώσουμε όλα τα κράτη-μέλη και τους λιμένους τους να εγκαταστήσουν νέα μηχανήματα, έτσι. Ε, η διαδικασία πώς έχει, εξετάζουμε προσεκτικά αυτές τις νέες τεχνολογίες και μετά τον Απρίλιο, μετά από τεκμηριωμένη ανάλυση, όπου θα έχουμε εξετάσει όλες τις πτυχές νέας τεχνολογίας, μετά θα υποβάλουμε πρόταση. Και εγώ έχω ενδιασμού σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα, όπω είπε ένα συνάδελφο για τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. Αλλά γιατί να τι απορρίψουμε εξ αρχή. Ε, προχωράει δυστυχώ η τρομοκρατία και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλε τι τεχνολογικέ εξελίξει και εμεί από πλευρά μα για να προασπίσουμε του ε, πολίτε μα. Ε, Α μην δαιμονοποιούμε τι νέε τεχνολογίε. Μαζί με την κυρία Μάνστρομ και την κυρία Ρέντινγκ θα προτείνουμε κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση με όλα τα προαπαιτούμενα για τα τεχνολογικά, νομικά ζητήματα, ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιωτικής ζωής. Όλες, όλες οι πτυχές θα καλυφθούν και θα προτείνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Χρειάζεται συνένεση για να έχουμε μία ευρωπαϊκή θέση και αυτό το αντιλαμβάνονται σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτό προβλέπεται να γίνει στο εγγύς μέλλον. Θα υποβάλουμε έκθεση. Τώρα συνεχίζουμε, συνεχίζουμε τις συζητήσεις και δεν υπάρχει συνωμοσία. Πιστέψτε με για να εγκαταστήσουμε πάρα αυτά νέα μηχανήματα και δεν υπάρχει στεγανή νέα τεχνολογία από πλευράς ασφαλείας. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα της ασφαλείας ασφάλεια. Χρειαζόμαστε κοινέ προσπάθειε, ε, μετά και ισχυρότατη διεθνή συνεργασία. Μετά από αυτή την έκθεση που θα υποβάλουμε θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσει ε, και θα προτείνουμε κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για να δούμε ποια θα είναι τα πρότυπα, ποιε θα είναι οι απαιτήσει, αν τα κράτη-μέλη επιλέξουν τελικά να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν νέε τεχνολογίε. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα. Η αντιτρομοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Έχουμε επώδυνε εμπειρίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη τρομοκρατία και τη απειλή όχι μόνο για τα άτομα αλλά και τι ίδιε κοινωνίε, τη δημοκρατία και τι θεμελιώδει μα αξίε. Ε, τα κράτη-μέλη φυσικά έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη και την ευθύνη ε, για τα συστήματα πληροφοριών του αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να συντονιστούμε και να ε, ε, χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα ζητήσω από τι υπηρεσίε μου ταχύτατα να κάνουν ανάλυση των πολιτικών του πλαισίου, των εργαλείων που ήδη έχουμε στη διάθεσή μα για να δούμε τι επιδέχεται βελτίωση και πώ μπορούμε ευφιέστερα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Και συμφωνώ με του συναδέλφου που είπαν και είμαι και εγώ πεπισμένη ότι η Europol, η Eurojust, οι εθνικέ αρχέ μπορούν να εργαστούν καλύτερα και με πιο συντονισμένο τρόπο και σίγουρα θα βρούμε μέτρα για να το καταφέρουμε αυτό. Στο Detroit αυτό που συνέβη και άλλα αντίστοιχα είναι σημαντικά διότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρομοκρατία και συνιστά σημαντικότατη απειλή ακόμη και πρέπει εμείς οι πολιτικοί να τα κινηθούμε ταχύτατα για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Αυτό είναι φυσιολογικό και επόμενο. Αλλά επίσης φέρουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε την ασφάλεια, ναι μεν, αλλά Αφού έχουμε κάνει διεξοδική ανάλυση και αξιολόγηση και ενδελεχή συζήτηση για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα, όπω είπε ο Επίτροπο Σιμ Κάλλα και όπω είπε και ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και πρέπει να λάβουμε υπόψη το πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι θα εργαστεί η Επιτροπή και θα επανέλθουμε με λεπτομερέστερε προτάσει αφού περατωθεί η αξιολόγηση και θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Σα ευχαριστούμε για αυτή την τόσο σημαντική ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κλείνει την ε, συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Και όσο μιλάτε, παρακαλώ και η Επιτροπή να αλλάζει για την επόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία. Δεν, ε, διαδικαστικό απλώ θα ήθελα να πω ότι εξεπλάγει. Γιατί στο, όταν βγήκε το ΚΑΘΙΑ, εγώ σήκωσα το χέρι μου και είχατε ήδη τον κατάλογο πλήρη. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε πώ θα γίνει αυτό, ποια είναι τα κριτήρια που δίνεται ο λόγο με το Α, Εγώ σήκωσα πρώτη το χέρι μου και εσύ είχατε κατάλογο. Ακριβώ τη στιγμή που εμφανίστηκε Eye σήκωσα εγώ το χέρι μου. Και εσεί ε, ήδη μα διαβάσατε ένα πλήρη κατάλογο. Θα ήθελα απλώ να εκφράσω την έκπληξή μου Πώ συνέβη αυτό και για μελλοντική χρήση να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Επιτρέψτε μου να σα εξηγήσω, εξηγήσω τη διαδικασία πολύ απλά από την στιγμή που αρχίζει μια συζήτηση έχει το δικαίωμα ένα μέλος να σηκώσει το χέρι του για το catch the eye που θα πει ότι εάν έρθετε προς το τέλος της συζήτησης και ζητήσετε το λόγο ενδέχεται να έχουν ήδη εγγραφεί πάρα πολλοί. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε 19 ανθρώπους εγγεγραμμένους και κανονικά έπρεπε να δώσω το λόγο μόνο για 5 λεπτά έκανα μία εξαίρεση και έδωσα από όλες τις ομάδες κάποιους αλλά δεν μπορούσα να πάρω και αυτού που είχαν μπει στο τέλο. Ζητώ συγγνώμη. Έχετε υπόψη από εδώ και πέρα ότι από την αρχή μια συζήτηση όποιο σηκώνει το χέρι καταγράφεται.